Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε στην συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για την χρηματοδοτική συνδρομή. Γίνεται απευθεία αναμετάδοση τη συνεδρίαση από το διαδίκτυο και θα ήθελα να ευχαριστήσω του επιτρόπου Μοσκοβισή και Νομπρόφσκη που είχαν την καλοσύνη να δεχτούν την πρόσκλησή μα και να έρθουν να μα ενημερώσουν για τη συμφωνία για το ελληνικό πρόγραμμα που υιοθετήθηκε στο Eurogroup της 24ης Μαΐου και που δεν έχει καταλήξει τεχνικά συμπεράσματα ακόμη, γιατί υπάρχουν ακόμη κάποιες εκκρεμότητες που συνεχίζουν να είναι αντικείμενο συζήτησης, αλλά ευελπιστούμε ότι θα καταλήξουμε σε αίσιο πέρας, ώστε να ολοκληρωθεί η τελική αξιολόγηση. Ήταν πολύ σημαντική η συμφωνία της 24ης Μαΐου, όχι γιατί ευελπιστούμε ότι θα... Θα οδηγήσει στην εκταμείευση της πρώτης δόσης από τα 10,3 δις για να πληρωθούν ε, τα λεξιπρόθεσμα και οι πιστωτές και επίσης θα ανοίξει το δρόμο για μια μεταγενέστερη συζήτηση και για την ελάφρυση του και για όλα αυτά μας ενδιαφέρουν οι απόψεις και η ενημέρωση των επιτρόπων. Προτείνω λοιπόν να δώσουμε αμέσω το λόγο στους επιτρόπους μας για να κάνουν εισαγωγικέ παρατηρήσεις 10 λεπτά συνολικά και μετά θα γίνει συζήτηση με τη διαδικασία του Catch the Eye. Πρώτα ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόφσκης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλησπέρα σας αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Όντως, όπως είπε και ο κύριος Γουαλτιέρη, πριν από δύο εβδομάδες το Eurogroup κατέληξε σε συμφωνία για την Ελλάδα. Μία συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για σημαντικές εκταμιεύσεις ποσών και επίσης εντοπίζει και ένα πακέτο για τα μέτρα του χρέους. Είναι το αποτέλεσμα πολύμινης αργόντως προσπάθειας και εργασιών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστά και αφοσιωμένα στήριξε και βοήθησε την όλη διαδικασία και μάλιστα μια συμφωνία σε επίπεδο προσωπικού ε, και η Βουλή των Ελλήνων υιοθέτησε ένα σημαντικό πακέτο μεταρρυθμίσεων, πολύ σημαντικό τέτοιο πακέτο μεταρρυθμίσεων και με βάση τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, χάρη στο πακέτο αυτό, θα μπορέσει η Ελλάδα να, φτάσει στο 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα μέχρι το 2018, που είναι ο βασικός στόχος και επίση επιτρέπει και το μηχανισμό προληπτικών μέτρων ή αυτόματη διόρθωσης για να βελτιωθεί η κατάσταση της οικονομίας. Και είναι τα βασικά στοιχεία αυτού του μεταρρυθμιστικού πακέτου. Βασικέ ε, μεταρρυθμίσει στη φορολογία και τι συντάξει, μέτρα για την εφαρμογή τη στρατηγική για να αντιμετωπιστούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ενίσχυση τη ανεξαρτησία ε, τη ε, διοίκησης για τα περιουσιακά στοιχεία, σύσταση νέου ταμείου αποκρατικοποίησεων και άνοιγμα αγορών ενέργειας. Ε, φυσικά συνεχίζονται και οι προσπάθειες ε, για την υλοποίηση των προαπαιτουμένων. Πάντως μπορούμε ήδη να διαπιστώσουμε σημαντική και αισθητή πρόοδο άρα βρισκόμαστε προς την ολοκλήρωση των προαπαιτουμένων Βέβαια η συμμόρφωση με όλα τα προαπαιτούμενα είναι η πρώτη προϋπόθεση για την εκταμείευση της πρώτης δόσης. Η δόση αφορά 10,3 δισεκατομμύρια ευρώ, διόλα μελιτέο ποσό, που θα καταβληθεί σε αρκετές δόσεις και θα επιτρέψει μία ικανοποίηση πολλών ληξιπρόθεσμων οφειλών και μία τακτοποίηση συσσωρευμένων τέτοιων ληξιπρόθεσμων ωφελών. Επίσης, ανοίξει το δρόμο για τη ε, υιοθέτηση κάποιων μέτρων για το χρέος, κάποια βραχυπρόθεσμα για τη διαχείριση του χρέους, προτεραιότητα και ε, προβλέπονται και μεσοπρόθεσμα μέτρα μετά την ε, ε, με την, με την ε, θετική υλοποίηση του προγράμματος ε, του Ταμείου Σταθερότητας, επίσης το θέμα της, των μη δανείων και αν παρεστεί ανάγκη και κάποια άλλα δάνεια, προφάλιγα άλλων δανείων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και πιο μακροπρόθεσμα, δηλαδή μετά το τέλος του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και ένας μηχανισμός αυτόματης διόρθωσης ή προληπτικών μέτρων που θα ενεργοποιηθεί από το Eurogroup σε περίπτωση που υλοποιηθεί ένα πιο δυσμενές σενάριο. Επίσης, ανάλογα με την, ε, και με βάση την θετική ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγηση και μετά από υιοθέτηση και των ε, μέτρων για το χρέο, θα ε, γίνουν και κάποιες ρυθμίσεις με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι μεταρρυθμίσει με βάση του προγράμματο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα. Θεωρούμε ότι οι μεταρρυθμίσει αυτέ θα επιτρέψουν την ανάκαμψη τη ελληνική οικονομία, την ανάκαμψη και την απόκτηση τη οικονομική σταθερότητα, μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση τη εμπιστοσύνη των επενδυτών αλλά και των πολιτών. Φυσικά, ε, ε, τα νομοσχέδια είναι ένα τμήμα τη προσπάθεια Αυτό που προέχει είναι η αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των μέτρων. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις ε, θα, θα πρέπει να γίνει ένας συντονισμό από την ε, Υπηρεσία Στήριξη των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και Φυσικά, βέβαια, στη τελική ανάλυση οι εθνικέ αρχές είναι αρμόδιες για την ε, έμπρακτη εφαρμογή. Υπάρχει τεχνική συνδρομή, όμω, σε όλου του βασικού τομεί μεταρρύθμιση με βάση το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα. Προβλέπεται συνδρομή για την εφαρμογή μέτρων που αφορούν την διοίκηση, ε, τη δικαιοσύνη, το επιχειρηματικό περιβάλλον ε, αποκρατικοποίησης, ε, υπηρεσίες υγείας και ούτω καθεξής. Εμπειρογνώμονες μας βρίσκονται ήδη επιτόπου, βοηθώντας την ελληνική διοίκηση για να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον με την απλούστευση της χορηγήση αδειών και βελτίωση της φορέ πρακτική ικανότητας. Περαιτέρω τεχνική συνδρομή ε, προβλέπεται και στην αγορά των σχέσεων, στην υγεία, τις μεταφορές και την πρόθεση των εξαγωγών. Επίσης είναι σημαντικό η Ελλάδα να αξιοποιήσει στο έπακρο τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια και γι' αυτό θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να επιταχύνουν το διοικητικό και το νομοθετικό έργο ώστε σχέδια ε, του, του, πακέτου 2017-2020 να ε, υλοποιηθούν και αυτό προϋποθέτει όλα τα προαπαιτούμενα για την περίοδο του 2014-2020 να αντικαταστηθούν από ένα, νομοθετικό, νομοθετικό πλαίσιο μέχρι τα τέλη του χρόνου. Τέλος, ε, ε, το πρώτο ε, επενδυτικό σχέδιο για επενδύσεις της Κρέτα Φαρμ έλαβε χρηματοδότηση από την ΕΤΕ με την υποστήριξη διαρθρωτικών επενδύσεων 15 εκατομμύρια είναι, μέρος, ε, είναι δάνειο της ΕΤΕ με εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Αυτό είναι το πρώτο σχέδιο, πολλά θα ακολουθήσουν για την Ελλάδα, πολύ σημαντικό αυτό το σχέδιο της Κρέτα Φάνους. Και εδώ θα βάλω τελεία και θα αφήσω τον Επίτροπο Μοσκοβισή για να σας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των προγραμμάτων. Ευχαριστώ, Επίτροπος Μοσκοβισή έχει το λόγο. Ευχαριστώ, ο Βάλτης έκανε μια γενικότερη παρουσίαση του προγράμματος. Εγώ θα προσπαθήσω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες τριών ε, στοιχείων. Πρώτον, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για τις ε, δόσεις. Δεύτερον, το θέμα του προληπτικού αυτού μηχανισμού. Και τρίτον, βεβαίω το θέμα της ε, υλοποίησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς η Ελλάδα μπορεί να παίρνει δύσκολες αποφάσεις. Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης θα δείξει κατά πόσον αυτή η ε, μεταρρύθμιση υλοποιείται. Όπως είπε και ο εξαιρετικός μας συνάδελφος ε, κύριος Σόιμπλε, όλα τελικά εξαρτώνται από την υλοποίηση implementation. Με αυτόν τον τρόπο θα ξεκινήσει η οικονομία και με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν νέες θέσεις τα νομοσχέδια λοιπόν πέρασαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, το θέμα το ασφαλιστικό και με ένα νομοσχέδιο στις 22 Μαΐου. Δύσκολα μέτρα σε μια πολύ σύντομη χρονική περίοδο πέρασαν από το ε, Κοινοβούλιο της Ελλάδας. Βλέπουμε όμως ότι ο έλεγχος θα ακολουθήσει ex για να δούμε κατά πόσο υλοποιούνται αυτά τα μέτρα. Το 95% των μεταρρυθμίσεων πέρασαν βεβαίως από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Όλα δεν έχουν ακόμα περάσει, αλλά είμαι σίγουρος ότι η Αθήνα θα κάνει αυτό που πρέπει, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν τα ε, λίγα σημεία τα οποία παραμένουν ακόμα ε, ανοιχτά και δεν έχουν περάσει από το Κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα ελπίζουμε να μπορέσει να ληφθεί η απόφαση για να ε, ελευθερωθεί το ποσό. Επαναλαμβάνω, η δόση αυτή 10,3 δις, ένα σημαντικό ποσό, θα επιτρέψει στην Ελλάδα να αντέξει 6 μήνες αυτό το μήνα, τον Ιούνιο, 7,2 δις 7,5 δις ε, ευρώ που θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να εξοφλήσει ε, κάποια λήξη πρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ε, ιδιώτες και βεβαίως ε, η συζήτηση όσον αφορά το υπόλοιπο κομμάτι της διαπραγμάτευσης, δηλαδή το θέμα του χρέους, θα ξεκινήσουν μετά το ε, τέλος του καλοκαιριού. Θα ξεκινήσει λοιπόν πρώτον η εξόφληση και κατόπιν θα ακολουθήσει με ένα δισεκατομμύριο αυτό που προβλέπεται από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού κράτους, η διακυβέρνηση και όλοι οι άλλοι τομείς οι οποίοι μέσω του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας πρέπει να καλυφθούν. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Επαναλαμβάνω, έχω εμπιστοσύνη σε ελληνικές αρχές και πιστεύω ότι θα προχωρήσει ε, τους ε, επόμενους μήνες και τις επόμενες μέρες το χρονοδιάγραμμα όπως έχει προβληθεί. Τώρα, το θέμα της αξιολόγησης και το θέμα ε, των προληπτικών μέτρων και του μηχανισμού αυτόματης διόρθωσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο για μας στην Επιτροπή, ε, ξέρετε πώς εκφραστήκαμε από αυτού, εμείς θεωρούμε ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι ικανά να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Όμως βάση του άρθρου 233 του πολυνομοσχεδίου προβλέπεται ένας τέτοιος προληπτικός μηχανισμός και ε, στο Eurogroup ε, αξιολογήθηκε αυτή η πρόταση. Πρόκειται για κάτι το οποίο με αντικειμενικό τρόπο θα αξιολογήσει αν ναι ή όχι ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα και αν υπάρχει ανάγκη αυτών των ε, προληπτικών μέτρων, αυτού του προληπτικού μηχανισμού. Ε, υπήρξαν κάποιες προηγούμενες εκτιμήσεις που ενδεχομένως ε, άφηναν να εννοηθεί ότι δεν πρόκειται για αυτόματο μηχανισμό. Όχι, πρόκειται για αυτόματο μηχανισμό και βεβαίως θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που οι στόχοι δεν υλοποιούνται. Το θέμα τώρα της βιωσιμότητας του χρέους, του ελληνικού χρέους, της 9 Μαΐου εκφράστηκαν οι υπουργοί επ' αυτού και βεβαίως αυτό γίνεται στις τρεις φάσεις, στη βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους. Οι πρώτες ανάγκες, 15% του ΑΕΠ τις τα πρώτα 15 χρόνια και μεγαλύτερο ποσοστό για τα επόμενα χρόνια. Η ιδέα, αν θέλετε, πίσω από αυτήν την ε, πρόταση είναι να υπάρχει μια σταθερότητα και μέχρι το 2018 ουσιαστικά γίνεται απλή διαχείριση χρέους. Από εκεί και πέρα, βάσει του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, η Ελλάδα θα πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Άρα, από το 2018 ε, θα ε, υπάρχει ανάγκη νέων μέτρων για το χρέος. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό όμως είναι ότι σήμερα και βλέπουμε αυτό από τη δήλωση του Eurogroup ότι είναι ξεκάθαρο από τις, τους υπολογισμούς των κρατών μελών πού θέλουμε να φτάσουμε. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να λάβουμε σήμερα μέτρα επί του χρέους ε, χωρίς σήμερα να υπάρξει καμία, αν θέλετε, ονομαστική μείωση αυτού του χρέους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες έτσι ώστε η Ελλάδα να ξαναβρει την εμπιστοσύνη των χρηματαγορών. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό και το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ. Η σημερινή κατάσταση είναι εξής. Το του δέχτηκε να κάνει την εξή σύσταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο πριν το τέλος του 2017 να παραμείνει το Δουνουτού την ε, στο ελληνικό πρόγραμμα εφόσον βεβαίως η ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους ε, είναι ικανοποιητική, θετική. Και αν κοιτάξουμε τα πράγματα με λίγη απόσταση, διαπιστώνουμε ότι πριν από ένα χρόνο ακριβώς μιλούσαμε για Brexit. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει πλέον στο σκηνικό. Εδώ και τέσσερα χρόνια συμμετέχω εγώ στο Eurogroup. Είμαι ένας από τους πιο παλιούς, να μην σας πω ο πιο παλιός, με το Μάριο Ντράγκη. Η ατμόσφαιρα έχει αλλάξει εντελώς. Και πλέον δεν μιλούμε για έξοδο διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα κάνει μεταρρυθμίσεις. Αυτό δεν έγινε βέβαια αυθόρμητα. Σήμερα όμως γίνονται μεταρρυθμίσεις και πρέπει να διασφαλίσουμε την υλοποίηση αυτών ε, που αποφασίζει η Ελλάδα. Και αυτό που είναι για μας σημαντικό σήμερα είναι να δούμε τις επενδύσεις. Οι αριθμοί που έχουν υποβληθεί σήμερα για μας είναι ρεαλιστικοί. 2,7 είναι η προβλεπόμενη ανάπτυξη του 2017. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εάν βεβαίως λειτουργήσει το σύνολο των μέτρων που ε, έχουν αποφασιστεί. Θέλουμε σε κάθε περίπτωση να στηρίξουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις και πιστεύω ότι θα είναι θετική απόφαση του Eurogroup όπως ακριβώς ε, πρότεινε η προηγούμενη συνάντηση. Ευχαριστώ. Όπως είπα, θα έχουμε συζήτηση με τη διαδικασία Catch the οπότε παρακαλώ ποιος θέλει το λόγο στο δηλώσει στη γραμματεία για να το σημειώσει. Θα ήθελα εγώ να θέσω τις πρώτες ερωτήσεις. Καταρχήν, να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ελληνική κυβέρνηση. Ναι, να το σημειώνουμε, το σημειώνουμε. Να σας ευχαριστήσω γιατί συμβάλλατε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ε, αίσια έκβαση του προγράμματος. Σε παρακολουθούν, τα σημειώνουν όλα, τα σημειώνουν κατά λεπτός. Μην ανησυχείτε, όλοι όσοι ζητάτε το λόγο θα τον λάβετε. Νομίζω ότι είναι πολύ θετική έκβαση και σε ό,τι αφορά την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης να δείξει ότι μπορεί να δρά, να αποκρίνεται και να επιλύει μείζονε κρίσει. Όπω είπατε, ότι το Brexit έχει φύγει από το πρόγραμμα, δεν είναι καν στον ορίζοντα και αυτό είναι πολύ θετικό. Έχω μια ερώτηση για τα μέτρα του χρέου. Καταρχήν, μέσο πρόθεσμα, πώ ερμηνεύεται αυτή το, αυτό το πιθανό δεύτερο πακέτο μέτρων. Τι θα πει πιθανό δεύτερο πακέτο μέτρων. Δηλαδή, αν παραστεί ανάγκη για την ε, ε, υλοποίηση των κριτηρίων αναφοράς και αν ε, υλοποιηθούν τα μέτρα θα γίνει αυτό. Με, είναι, ότι είναι πιθανό και δεύτερο πακέτο μέτρων. Με, αυτό το, με αυτή την ερμηνεία είναι δυνατό ή υπάρχει κάτι άλλο. Ή δεν είναι σαφές δηλαδή ακόμη ότι αν υλοποιηθούν αυτοί οι δύο όροι θα υπάρχει και δεύτερο πακέτο. Σε ό,τι αφορά τον μηχανισμό αυτόματης διόρθωσης για το χρέος, είναι κάτι που αφορά το μακροπρόθεσμο ορίζοντα και αυτός ο μηχανισμός είναι πολύ θετική πρόταση. Βέβαια, το 5% των θεμάτων ακόμη εκρεμή. Και τι γίνεται με την επιστροφή του, του ΕΚΑΣ. Έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα για την καταβολή του ΕΚΑΣ. Καταρχήν, να απαντήσω εγώ για το θέμα αυτό χωρίς να επισέλθω σε υπερβολικές λεπτομέρειες, γιατί μιλούμε για συζήτηση που άπτεται της ε, ομάδας εργασίας του Eurogroup, που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί. Όταν είπα 5% ήταν ε, κατά προσέγγιση, μπορεί να είναι 2%, μπορεί να είναι 7%, ε, ενώ ότι υπάρχουν ακόμη κάποιοι περιορισμοί από τα κρατη και ότι δεν υπάρχει ακόμη τυπική επίσημη συμφωνία για το πακέτο. Πάντως αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι το Euro Working Group ε, γενικώ συμφωνεί. Υπάρχουν εκκρεμότητες για ίσονο σημασία ζητήματα. Και στις συζητήσεις τις δύο τελευταίες εβδομάδες διαπίστωσα θεαματική πρόοδο προς την κατεύθυνση της συμφωνίας. Πάντως ε, πιστεύω ότι οι λίγες εκκρεμότητες θα διαθετηθούν όσο νοπό, ώστε να ληφθεί απόφαση στις 16 Μαΐου στο Eurogroup ε, η απόφαση για την εκταμίευση. Συνεχίζεται η πρόοδος και εγώ είμαι αισιόδοξο ότι θα ληφθεί η συμφωνία. Τώρα για τα μέτρα και οι δύο ερμηνείες είναι Να σας δώσω τη δική μου ερμηνεία και με τον κύριο Ντομπρόφσκη συμμετέχουμε στις ίδιες συνεδριάσεις, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι μέχρι το 2018 θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη διαχείριση του χρέους. Και εκεί έχουμε δύο κόκκινες γραμμές που είναι σαφείς. Η πρώτη κόκκινη γραμμή είναι ότι κανείς δεν θέλει να επανέλθει στο θέμα του προγράμματος και δεύτερον ότι κανείς δεν είναι υπέρ οποιοδήποτε κουρέματος Τώρα, μετά το τέλος του προγράμματος, το 2018, υπάρχει πιθανότητα να χρειαστούν πιο φιλόδοξα μέτρα για το χρέος, αλλά μπορεί να είναι και αφίδρομα. δηλαδή μπορεί να μην υπαραστεί ανάγκη για τέτοια μέτρα νέα. Βέβαια όλοι γνωρίζουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστούν. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι είναι δυνατό και αυτό να το καθορίσουμε μέχρι τα τέλη του έτους. Δηλαδή τι μπορεί να γίνει εκεί. Αυτά. Και ίσως ο κύριος Ντομπρόφσκης ε, θέλει να προσθέσει κάτι. Yeah, maybe <clears throat> just to uh, Να αναπροσθέσω κάτι, ένα σημείο σε αυτά που είπε ο Πιέρ. Σε κάθε περίπτωση στο δεύτερο εξάμεινο του έτους θα επανέλθουμε στο θέμα του χρέους, γιατί εκεί θα πρέπει να κρυθεί η συμμετοχή ή όχι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα. Μετά λοιπόν την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και μετά όσον αφορά, μετά την συμφωνία, συγγνώμη, όσον αφορά τα μέτρα για το χρέος, εκεί θα πρέπει να ξαναδούμε το πρόγραμμα, δηλαδή θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες και θα ξανασυζητήσουμε το θέμα του χρέους το δεύτερο εξάμεινο του έτους και βεβαίως αυτό είναι και αποτέλεσμα της ε, ανάλυσης βιωσιμότητας του χρέους. Ο Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση που θα ήθελα να κάνω στον Αντιπρόεδρο Ντομπόφσκης και στον Επίτροπο Μοσκοβισή. Στις 30 Μαΐου, δηλαδή πριν από λίγες μέρες, η αρχή, η στατιστική αρχή της Ελλάδας έδωσε τα στοιχεία για το πρώτο τριήμινο του 2016. Και αυτό που το, μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε στοιχεία για το ΑΕΠ, και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μία μείωση τάξης του 0,5%. Και αυτό βεβαίως συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία και την ε, Τράπεζα της Ελλάδας. Μιλάμε λοιπόν ε, για μία κατάσταση η οποία μας ε, οδηγεί αν θέλετε, σε κάποια ερωτηματικά. Το 2015 είχαμε προαναγγείλει μια πιο αισιόδοξη κατάσταση και μια επιστροφή στην ανάπτυξη. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πώς εκλαμβάνετε αυτούς τους αριθμούς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Σε ό,τι αφορά τα μακροοικονομικά δεδομένα, οι προβλέψεις ε, για το πρόγραμμα όταν έγινε η συμφωνία για το πρόγραμμα ήταν 0,5 ύφεση πέρυσι και 0,3 φέτος ύφεση. Τελικά ε, για πέρυσι ήταν 0,2 καλύτερα από τις προβλέψεις η ύφεση, ήταν λίγο λιγότερη και για φέτος οι προβλέψεις ε, των θεσμών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι το πρώτο εξάμεινο θα συνεχιστεί η ύφεση και μετά θα επιστρέψουμε στην πορεία της οικονομικής ανάπτυξης κατά το δεύτερο εξάμεινο του έτους. Με συνολικό όμως ποσοστό 0,6, δηλαδή αρνητική ανάπτυξη. Οπότε τα δεδομένα αφορούν περισσότερο τις πιο αρνητικές προβλέψεις, αλλά προς το παρόν δεν εξασφαλίζουν αναθεώρηση, δεν δικαιολογούν αναθεώρηση των προβλέψεων, των νεαρινών προβλέψεών μας. Και ένας από τους λόγους είναι και η καθυστέρηση της πρώτης αξιολόγησης. Γιατί εξαιτία αυτής της καθυστέρησης παρατάθηκε και η αβεβαιότητα η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης ε, είναι σημαντικό μήνυμα και προς τους ε, επενδυτές και προς τους πολίτες ότι η Ελλάδα ξαναμπαίνει στον καλό δρόμο και εξασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα που είναι και προαπαιτούμενο, απαραίτητη προϋπόθεση μάλλον για την οικονομική ανάπτυξη. Υπερβάνος Μπερές. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους δύο επιτρόπους. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά αυτά τα μέτρα, το, τα προληπτικά, το μηχανισμό αυτό με τις διόρθωσεις. Ε, από ό,τι ξέρω τα υιοθέτησε η Βουλή των Ελλήνων. Με βάση όμως ποιους κανόνες προτάθηκαν αυτά τα μέτρα του, το μηχανισμού προληπτικών μέτρων και φοβάμαι πως αποτελέσουν πια βασικό τμήμα της ε, και των υπόλοιπων προγραμμάτων που θα υποβληθούν ε, σε άλλες χώρες. Δηλαδή μήπως χρησιμοποιηθεί η Ελλάδα προηγούμενο για να απαιτούνται τέτοια μέτρα και τέτοιο μηχανισμός προληπτικό μέτρο και από άλλες χώρες. Από ό,τι ξέρω, τέτοιο μηχανισμό προληπτικό μέτρο στερείται νομικής βάσης. Τώρα, δεύτερη ερώτηση για το χρέος. Όλοι χαιρόμαστε που το θέμα του χρέου βρίσκεται επιτάπητο και έγιναν κάποιε συζητήσεις σχετικά. Πάντως ε, οι σημερινές συνθήκες ε, ε, αποπληρωμής του χρέους ανησυχούν ιδιαίτερα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, ποιος τελικά ευνοείται από αυτές τις ρυθμίσεις. Και εσείς μας μίλησατε για το χρονικό ορίζοντα του 2018. Ε, μήπως υπάρχουν όμως επιχειρήματα για να διαψεύσουμε αυτούς που λένε ότι όλες οι ρυθμίσεις του χρέους γίνονται για να μπορέσει η Ελλάδα ουσιαστικά να αποπληρώσει τα χρέη της στις δικές μας τράπεζες. Και άρα δεν θα ωφελήσουν άμεσα τον ελληνικό κορβανά. Ναι, όσον αφορά αυτό το προληπτικό μηχανισμό, κοιτάξτε, πρόκειται για μια λογική που έχει εμφανιστεί και άλλες φορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί από την αρχή ότι αυτός ο μηχανισμός δεν ήταν απαραίτητος. Απολύτως απαραίτητος δεν ήταν σύμφωνα με τους δικούς μας υπολογισμούς. Διότι, επαναλαμβάνω, τα μέτρα που ελήφθησαν κανονικά αρκούν και επαρκούν για να φτάσουμε στα ποσοστά ε, τελικά, δηλαδή, ήμασταν μάλλον αντίθετοι. Τελικά όμως συμφωνήθηκε ότι αυτός ο προληπτικός μηχανισμός ε, έπρεπε να υιοθετηθεί και βεβαίως από εκεί και πέρα η κάθε κυβέρνηση αποφασίζει ποια θα είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που θα πάρει τα τρία επόμενα έτη για να υλοποιηθούν αυτές οι αποφάσεις. Ο αυτόματος μηχανισμός όμως αυτός, ε, όπως καταλαβαίνετε, ενεργοποιείται στην περίπτωση που δεν τηρηθούν αυτοί οι στόχοι. Νομίζω λοιπόν ότι δεν είναι κάτι που ευσταθεί η ανησυχία σας όσον αφορά το δημοκρατικό έρισμα αυτών των ε, μέτρων και αυτού του μηχανισμού. Ε, όσον αφορά τώρα το δεύτερο ερώτημά σας, αρχικά πρέπει να σας πω ότι ήμασταν ε, υπέρ μιας συνολικής συμφωνίας, μιας συμφωνίας επί της αρχής που δεν είναι βραχυπρόθεσμη. Δηλαδή, μέχρι το 2018, μετά δεύτερη μεσοπρόθεσμη φάση μέχρι το τέλος του προγράμματος και επέκεινα. Ο Βάλτης του είπε πολύ σωστά ότι εδώ θα πρέπει να υπάρχει μια συνολική αντιμετώπιση. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο. Εγώ ήθελα να κάνω... Εγώ ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Για το θέμα του χρέους, φαντάζομαι ότι ξεκινώντας κανείς να ρυθμίσει το θέμα του χρέους, θα πρέπει να στηριχθεί στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ο κανονισμός 472 του 2013, που στο άρθρο 7, παράγραφος 9, λέει ότι το κράτος μέλος εξετάζει τους λόγους για τους οποίους έχει φτάσει το χρέος σε αυτό το ύψο και ενδεχόμενα αν υπάρχουν παρατυπίες. Δεν βλέπω ούτε η Ελλάδα αλλά ούτε κι εσείς ως Κομισιόν να αξιοποιείτε αυτό τον κανονισμό. Το δεύτερο είναι γιατί δεν χρησιμοποιείτε την ε, μορφή με την οποία ρυθμίστηκε το χρέος για την Ουκρανία. Δηλαδή ένα haircut της τάξης του 20% και εξόφληση με ρήτρα ανάπτυξη, που σημαίνει ότι θα μπορέσει πραγματικά να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του χρέους και στο θέμα της ανάπτυξης. Πώς μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη όταν έχουμε την ίδια μέθοδο, την ίδια συνταγή, αυξημένους φόρους, φορομπηκτική πολιτική, δημοσιονομική προσαρμογή βίαιη και ενώ έχετε τώρα την ευκαιρία να αξιοποιήσετε κεφάλαια, όχι εσείς η Ελλάδα. Πρώτον, τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι οι επιστροφές των κερδών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των κεντρικών τραπεζών της Ευρωζώνης, S&P και ANFAS. Είχε πει ο κύριος Ντράγκη ότι μετά τη λήξη της αξιολόγησης αυτά τα ποσά είναι στη διάθεση της χώρας. Τώρα αυτά το Eurogroup τα κρατά για ενδεχόμενη μελλοντική χρηματοδότηση της Ελλάδας. Και δεύτερον, υπάρχει ένα περίσσευμα 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το δάνειο το τρίτο. Αυτά τα λεφτά, αντί να πέσουν είτε στην ανάπτυξη, είτε να ρυθμίσουν το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης του ασφαλιστικού συστήματος ή των κόκκινων δανείων, τα κρατάει το σύστημα, το ESM, για να τα χρησιμοποιήσει, για να δώσει χρήματα στα κράτη-μέλη, τα οποία ενδεχόμενα να ζημιωθούν από μια ρύθμιση του πρώτου δανείου, δηλαδή από μια επιμήκυνση και μια μελλοντική ίσως μείωση επιτοκίων. Τελικά δεν βλέπετε ότι τώρα υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία και στο θέμα του χρέους να κάνουμε μια κατεύθυνση σαν για αυτή που σας προτείνουμε, όπως επίσης και να αξιοποιηθούν τα κεφάλαια 10 δισεκατομμύρια ευρώ από την επιστροφή των χρημάτων των κερδών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα S&P και τα ΑΝΦΑΣ. Ευχαριστώ. Uh, Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας για το χρέος. Όντως το επίπεδο του ελληνικού χρέους είναι πολύ υψηλό, σχεδόν 180% του ΑΕΠ. Γι' αυτό και τα μέτρα για το χρέος είναι τμήμα της συζήτηση. Τώρα, αν δούμε το θέμα του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους, είναι εξωσημείωτο ότι τα δάνεια του Eurogroup της Ευρωζώνης που δόθηκαν στην Ελλάδα μέχρι, μέσω του μηχανισμού σταθερότητας ή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ε, δίνονται με πολύ ευνοϊκούς όρους, δηλαδή με πολύ χαμηλά επιτόκια, με μακρά περίοδο ρήμασης, με περίοδο χάριτος ε, και για το κεφάλαιο και για τους τόκους, με αποτέλεσμα οι το, κόστος καθαρής του, το καθαρό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους για την Ελλάδα ως τμήμα του ΑΕΠ είναι μικρότερο από ό,τι για άλλες χώρες όπως η Ιταλία ή η Πορτογαλία που έχουν υψηλότερο καθαρό κόστος ε, εξυπηρέτησης χρέους γιατί η Ελλάδα λαμβάνει δάνεια με πολύ ευνοϊκότερους όρους από τις υπόλοιπες χώρες. Τώρα, ποια είναι τα επόμενα βήματα. Αν κατάλαβα καλά, αναφερθήκατε στα κέρδη SMB και ΑΜΦΑ. Όντως ε, υπήρχε συμφωνία ως τμήμα του δεύτερου προγράμματος και μετά την ε, αίσια διεκπεραίωση του δεύτερου προγράμματος, τα κέρδη αυτά ή τα ισοδύναμα αυτών των κερδών θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Και μια και δεν ε, διεκπαιρεώθηκε θετικά ουδέποτε το δεύτερο πρόγραμμα, δεν ισχύει πια αυτή η συμφωνία. Τα συμπεράσματα του Eurogroup βέβαια επανέφεραν αυτό το θέμα στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Οπότε είναι κάτι που εξετάζεται στο Eurogroup ως ε, μεσοπρόθεσμο μέτρο για το χρέος. Οπότε έχει επανέλθει ε, στις συζητήσεις και αυτό το θέμα της επιστροφής των κερδών. θα απέφευγα συγκρίσεις ε, με την Ουκρανία γιατί η Ελλάδα έχει επωφεληθεί από πολύ μεγαλύτερη ανάμιξη του ιδιωτικού τομέα στη μείωση του χρέους από ότι η Ουκρανία. Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διέγραψε καθόλου από το επίσημο χρέος. Απλώς παρέχει χρηματοπιστωτική συνδρομή και το ε, μέγεθος της, του προγράμματος μακροχρηματοδοτικής συνδρομής για την Ουκρανία ήταν πολύ μικρότερο από ότι το αντίστοιχο πρόγραμμα για την Ελλάδα. Το τρέχον πρόγραμμα για την Ουκρανία είναι 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τα 86 δισεκατομμύρια ευρώ του τρίτου προγράμματος για την Ελλάδα και ε, ας προσθέσουμε και τα άλλα, βλέπετε ότι οι τάξεις είναι πολύ διαφορετικές. Ευχαριστώ. Okay. Ε, ε, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που είστε πάλι σήμερα μαζί μας. Εγώ είμαι αισιόδοξη από τη φύση μου. Θα προσπαθήσω λοιπόν, ακόμα και σε αυτήν εδώ την ε, ομάδα εργασίας, να παραμείνω αισιόδοξη. Και θεωρώ ότι είναι καλό το ότι εδώ μιλούμε για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και όχι μόνο για την υιοθέτησή τους αλλά και για την υλοποίηση, την εφαρμογή τους. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι είναι για σας ε, το νόημα της λέξης implementing. Εννοείται πλήρη εφαρμογή, μερική εφαρμογή, καλή εφαρμογή, ελλειπής εφαρμογή. Ποια είναι, ε, αν θέλετε, η έννοια της υλοποίησης και της εφαρμογής για σας όταν φτάσουμε σε ποιο επίπεδο και θα ήθελα ο Επίτροπος Μοσκοβισή να μου πει κάτι παραπάνω όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση της αποκρατικοποίησης. Ε, μιλήσατε για το χρονοδιάγραμμα. Μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω όσον αφορά τη λεπτομέρεια αυτού του χρονοδιαγράμματος. Κοιτάξτε, οι δύο σας ερωτήσεις είναι αλληλένδετος σαφώς και εγώ είμαι αισιόδοξο. γιατί πιστεύω ότι έχουμε προχωρήσει πολύ και έχει γίνει μεγάλη πρόοδος. Πριν από ένα χρόνο μιλούσαμε για Brexit. Σήμερα αυτή η προοπτική πλέον έχει εξαλειφθεί και οι μεταρρυθμίσεις ε, έχουν σχεδόν ε, όλες περάσει από το ελληνικό κοινοβούλιο, έχουν ψηφιστεί. Πιστεύω λοιπόν ότι ξεπεράσαμε σε μεγάλο βαθμό αυτήν την κρίση. Όταν μιλάμε λοιπόν για implementation, για υλοποίηση, βεβαίως και υπάρχουν διαρθρωτικά προβλήματα και δυσκολίες στην Ελλάδα όσον αφορά παραδείγματο χάρη την υλοποίηση αυτών που ψηφίζονται. Και σίγουρα κάποια από τα μέτρα που έχουν προωθηθεί είναι κάτι που έχει σαν σκοπό την καλύτερη υλοποίηση. Παραδείγματο χάρη, η Γενική Γραμματεία ε, Εσόδων. Αυτό είναι κάτι που σαφώς και εμπεριέχει και ένα στοιχείο παρακολούθησης της υλοποίησης ε, η δημιουργία ανεξάρτητης αρχής. Ε, όταν μιλάμε λοιπόν για υλοποίηση εννοούμε πλήρη υλοποίηση. Και όταν αναφέρεστε στα ποσά της ιδιωτικοποίησης. 15 δις, 15 δις και βεβαίως αυτό το ποσό θα πρέπει να ελεγχθεί. Αυτό είναι αυτό που περιμένουμε. Η πρώτη εκταμίευση, αυτά τα 7,5 δις, βεβαίως και έχουν σαν σκοπό να αποπληρωθούν τα ποσά που πρέπει να αποπληρώσει τον Ιούνιο η Ελλάδα και κατόπιν να καλυφθούν κάποιες ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημόσιου τομέα. Και βεβαίως το επόμενο ποσό, τα 2,5 δις, είναι κάτι που περιμένουμε να δοθεί πριν το τέλος του χρόνου και αυτό συγκρινόμενο με το ποσό του 2015 βεβαίως είναι πολύ χαμηλότερο. Όταν μιλάμε τώρα για την ιδιωτικοποίηση, την αποκρατικοποίηση. Βεβαίω και υπάρχει μια σχέση μεταξύ της ε, υλοποίηση ε, αυτών ε, για το οποίο έχει δεσμευθεί η Ελλάδα σε αυτό το τομέα και της εκταμίευσης των τόσων. Αλλά επαναλαμβάνω, όταν μιλάμε για implementation εννοούμε πλήρη υλοποίηση. Ο κύριος Παπαδημούλης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ντομπρόψης και κύριε Μοσκοβισή, σήμερα μας είπατε αρκετά θετικά νέα. Πρώτον, ότι είσαστε σίγουροι ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες λίγες μέρες και τυπικά η πρώτη αξιολόγηση. Σημειώνω ότι έχει να ολοκληρωθεί αξιολόγηση ελληνικού προγράμματος δύο ολόκληρα χρόνια, από την άνοιξη του 2014. Δεύτερον, ότι μέσα στον Ιούνιο θα δοθεί η δόση των 7,5 δις. Τρίτον, ότι πιστεύετε ότι το τρίτο πρόγραμμα για την Ελλάδα θα είναι και το τελευταίο και τέταρτον ότι έσπασε το ταμπού και όλοι πια δέχονται ότι πρέπει και οι δανειστές να κάνουν κάτι από την πλευρά τους για να καταστεί το ελληνικό δημόσιο χρέος βιώσιμο. Επειδή όμως ο ελληνικός λαός έχει υποφέρει πάρα πολύ για έξι χρόνια, με μια τεράστια ύφεση, με μια τεράστια δυσπιστία και είναι και αρκετά δύσπιστος απέναντι και στις καλές ειδήσει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πρώτα απ' όλα, μέσα σε αυτό το δεύτερο εξάμεινο που θα εξετάσετε πιο συγκεκριμένα, οι δανειστές, τα μέτρα που πρέπει εσείς από την πλευρά σας να πάρετε για να γίνει το ελληνικό δημόσιο χρέος βιώσιμα, ποια θα είναι, εξετάζετε το ενδεχόμενο πρόορης αγοράς των δανείων του IMF από τον ESM, όπως έχει ήδη προταθεί από τον κύριο Ρέκλινγκ, με αξιοποίηση του ποσού του προγράμματος που είναι 15 με 20 δες που δεν χρησιμοποιήθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έτσι ώστε να μειωθεί το επιτόκιο αυτού του δανεισμού. Όπως δεχτήκατε και ζητήσατε από την Ελλάδα αυτόν τον αυτόματο μηχανισμό εξισορρόπησης παρότι είπατε ότι κατά τη γνώμη σας μάλλον δεν χρειάζεται γιατί τα μέτρα θα αποδώσουν. Προκειμένου να ικανοποιήσετε την απέτηση του IMF. Τώρα που το IMF για να μείνει στο πιλωτήριο του προγράμματος ζητάει μια μεγάλη ελάφρυνση του χρέους. Η Κομισιόν τι θέση θα πάρει. Ξέρω ότι η αρμοδιότητα ανήκει στο ε, Eurogroup, αλλά εσείς ως Κομισιόν τι πιστεύετε. Και επίση, στην Ελλάδα οι πάντες, και η κυβέρνηση Τσίπρα και η αξιωματική αντιπολίτευση και ο κύριος Τουρνάρας, διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδας και πρώην Υπουργός Οικονομικών, λένε ότι χρειάζεται ρεαλιστικότερα, χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα από το 2018 και μετά έτσι ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή της Ελλάδας στην ανάπτυξη με επενδύσεις και μείωση της ανεργίας. Ποια είναι η θέση της Κομισιόν απέναντι σε αυτή την ιδέα. Uh, okay, quite a few... Αρκετές ερωτήσεις ε, υποβάλλεται. Ε, καταρχήν, αν κατάλαβα καλά, η πρώτη δόση του προγράμματος αυτού καταβλήθηκε ήδη τον Αύγουστο, πέρυσι. Πέρυσι τον Αύγουστο. Οπότε τώρα μιλούμε για τη δεύτερη δόση ουσιαστικά αυτού του προγράμματος. Και αν όλα βγουν καλώς, ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση στις επόμενες μέρες για να εκταμιευθεί και η επόμενη δόση τις ε, επόμενες εβδομάδες. Όπως είπα, η δόση αφορά 10,3 δισεκατομμύρια ευρώ και το πρώτο τμήμα, η πρώτη δόση θα είναι 7,5 δισεκατομμύρια που θα καταβληθούν αμέσως και στη συνέχεια θα έχουμε μερικές μικρότερες δόσεις που αφορούν την τακτοποίηση των λεξιπρόθεσμων οφειλών ή περίμερες οφειλές προς τον ιδιωτικό ληξιπρόθεσμο οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα. Θα δοθούν κάποια κονδύλια για το θέμα αυτό και είπατε ότι μιλήσατε για την πρόορια αγορά των δανείων του Δουνουτού και αντικατάστασή τους από δάνεια με ε, πιο χαμηλό επιτόκια. Αυτό όντως συζητήθηκε και μάλιστα αν διαβάσετε συμπεράσματα του Eurogroup για την ε, διαχείριση των φυλών, οποιαδήποτε ε, μερική ε, ε, πληρωμή από, από, δάνει, από δάνεια από μη χρησιμοποιούμενα κολλή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Αυτό όντως είναι ένα από τα μέτρα που μεσοπρόθεσμα συζητήθηκαν και συζητούνται και αυτά τα θέματα των δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου γιατί αφορούν υπάρχοντα επίσημα δάνεια. Τώρα, για τις μεικτές χρηματοδοτικές ανάγκες, ε, πρόθεση είναι οι αρχικές μεικτές χρηματοδοτικές ανάγκες να μην υπερβούν το 15% του ΑΕΠ και αργότερα να μην υπερβούν το 20% του ΑΕΠ. Και ανάγκη θα γίνει και επιπλέον reprofiling του χρέους σε ό,τι αφορά το στόχο του πρωτογενούς ε, πλεονάσματος. Δεν είναι πρόθεση των ε, δανειστών αυτό το 3,5% πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα, ε, πρωτογενές πλεόνασμα του ΕΠ για όλη την περίοδο ε, μέτρησης μέχρι το 2016 να μειωθεί σταδιακά στο μέτρο που και το δημόσιο χρέος ακολουθεί την πορεία που είχαμε προδιαγράψει. Σας ευχαριστώ. Ο Φίλιπ Λάμπερτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις και θα ήθελα να μου απαντήσουν και οι δύο ε, επίτροποι. Θα τις θέσω μία στα αγγλικά και μία στα γαλλικά. Είναι και για τους δύο. Συνεχίζοντας αυτά που είπατε κύριε Αντιπρόεδρε Ντομπρόφσκης. Είναι, είναι σαφέ και προφανέ ότι το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο δεν πιστεύει ότι είναι βιώσιμο το πρωτογενέ πλεόνασμα του 3,5%. Μίλησε για 1,5% πρωτογενέ ε, πλεόνασμα. Είπατε ότι θα μειώσουμε το χάσμα μέχρι τα τέλη του χρόνου και τι διαφορέ μα με το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Γι' αυτό τι σημαίνει ότι οι πιστωτέ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναθεωρήσουν και θα μειώσουν αυτό το πρωτογενέ ε, πλεόνασμα όχι για το 2060, αλλά πολύ νωρίτερα. Η δεύτερη ερώτηση. Αν ήσασταν και οι δύο ακόμα Υπουργοί Οικονομικών των αντίστοιχων χωρών σας, σήμερα, θα δεχόσασταν αυτό το προληπτικό μηχανισμό που επιβάλλεται σήμερα στην Ελλάδα. Πείτε μου ναι ή όχι και για ποιους λόγους. Στην πρώτη ερώτησή σας πιστεύω ότι οι αξιολογήσεις διαφέρουν σήμερα. Οι εκτιμήσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου διαφέρουν σήμερα. Γι' αυτό και δεν έχει νόημα να σας δώσω απάντηση. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θεωρεί ότι αυτό το 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα είναι υπερβολικό. Ναι, γιατί, γιατί θεωρούν ότι Ενάμιση είναι το πλεόνασμα αυτό και αυτό το ενάμιση πλεόνασμα το οποίο ουσιαστικά θα γίνει 5,5% πλεόνασμα σύμφωνα με τους δικούς μας κανόνες υπολογισμού. Ε, γι' αυτό και μέχρι το τέλος του χρόνου θα συζητήσουμε, θα επαξεργαστούμε αυτό το θέμα έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια κοινή ανάλυση ποιοσιμότητας του χρέους. Γι' αυτό και λέμε εξάλλου στα συμπαράσματα του Eurogroup ότι θα συνεργαστούμε στενά. Η απόφαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι ότι θα προτείνουν θετική ε, απάντηση στο ερώτημα αν ή όχι θα παραμείνουν στο ελληνικό πρόγραμμα. Και ελπίζουμε ότι αυτό ε, θα υιοθετηθεί σαν απόφαση και αυτό βεβαίως ε, μακροπρόθεσμα θα συνεχιστεί. Τώρα, το θέμα της βιωσιμότητας του χρέους είναι αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει από εδώ και πέρα τους επόμενους μήνες. Η δεύτερη ερώτησή σας, μα αυτό είναι κάτι που μου θυμίζει τηλεοπτικό παιχνίδι. Δεν είμαι υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας. Και επίσης θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας και το ίδιο ισχύει και τη χώρα του Βάλτης. Η Γαλλία δεν είναι, δεν ήταν και δεν θα είναι ποτέ πιστεύω μια χώρα η οποία θα βρίσκεται σε πρόγραμμα προσαρμογής και είμαι σίγουρος ότι οι Γάλλοι που συνήθως κλαίγονται και διαμαρτύρονται σε καμία περίπτωση, σε καμία δεν βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Μα θα δεχόσασταν ένα τέτοιο μηχανισμό για να παραμείνει η Γαλλία. Κοιτάξτε, έχουμε μηχανισμούς δημοσιονομικής προσαρμογής που δεν διαφέρουν και τόσο πολύ. Όταν υπάρχουν συστάσεις, χρονοδιαγράμματα και υποχρεώσεις και προσπάθειες διαρθρωτικές για μια χώρα, οι μηχανισμοί είναι αυτόματοι και πρέπει να είναι αξιόπιστοι. Και αφού μου κάνετε αυτή την ερώτηση και αναφέρεστε σε μια συγκεκριμένη χώρα, θέλω να σας πω ότι αυτό που λέει η Επιτροπή για τη Γαλλία, το λέει και το επαναλαμβάνει, ότι πρέπει να είμαστε κάτω από το 3% του ΑΕΠ, όσον αφορά το χρέος μας, και η Γαλλία έχει δεσμευθεί ότι θα το τηρήσει ο προαιρετικός μηχανισμός πρέπει να είναι προαιρετικός και πρέπει να είναι προληπτικός. Δηλαδή δεν πρέπει ε, να υπάρχει παρά μόνο για να μην χρησιμοποιείται υποκανονικά συνθήκας. Σας ευχαριστώ. Ο Μάρκος Φέρμπερ. Oh, Αν μήπως θέλετε να προσθέσετε κάτι. Τον Πρόφσκης. Και εγώ έχω ένα σχόλιο. Ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση. Κάτι που τόνισα και εγώ και ο Πιέρ. Το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο φαίνεται να έχει πιο απεσιόδοξε μακροοικονομικέ προβλέψει και επίση πιο απεσιόδοξη εκτίμηση της αποδοτικότητας των μέτρων που θα εφαρμόσει η Ελλάδα. Αν δείτε μέχρι στιγμής όμως το πρόγραμμα, πέρυσι ο στόχος ισοζυγίου ε, ε, ήταν πρωτογενές πλεόνασμα 0,5% και ε, χωρίς να λάβουμε υπόψη την ανακεφαλοποίηση ήταν 0,7 πρωτογενές πλεόνασμα. Σαφώς καλύτερη ε, σαφώς καλύτερο αποτέλεσμα από το προβλεπόμενο. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι με την εφαρμογή των παραμετρικών μέτρων ε, σε ύψο 6% του ΕΠΟ, όπω συνομοθέτησε η Ελλάδα, θα μπορέσουμε να περάσουμε από το 0,7% ε, ε, πρωτογενέ πλεόνασμα στο 1,5%. Ιδιαίτερα σε κατάσταση οικονομικής ανάπτυξης. Και αυτό αναμένεται ότι στο δεύτερο εξάμεινο του έτους η Ελλάδα θα επιστρέψει στο δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης. Τώρα, ήμουν υπουργό Οικονομικών πολύ καιρό πριν και την ένταξη κάτι που ήταν διαφορετικό. Και μάλιστα ήμουν και πρωθυπουργό κατά το πρόγραμμα της Λετωνίας, γιατί η Λετωνία είχε μνημόνιο. Και η στρατηγική που θετήσαμε ήταν να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να έχουμε εμπροστοβαρή προσαρμογή δημοσιονομική και στα πλαίσια των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για να ανακτήσουμε γρήγορα την ε, χρηματοπιστωτική μας σταθερότητα και έτσι να επιστρέψουμε ε, γρήγορα στο δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης. Και μάλιστα υιοθετήσαμε τα περισσότερα μέτρα στα μέσα του 2009. Και στο δεύτερο ήδη εξάμεινο του 2010 είχαμε επιστρέψει στην οικονομική ανάπτυξη. Και μάλιστα αμέσω μετά είχαμε από του ταχύτερου ρυθμού οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Οπότε, αν μπορώ να αντιλήσω κάτι από την προσωπική μου εμπειρία, είναι ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν τα απαραίτητα μέτρα για να ανακτηθεί η ε, χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική σταθερότητα το συντομότερο δυνατό. Ο Ούντο Μπούλμαν. Μάρκο Φέρμπερ. όχι λάθο, ο Μάρκο Φέρμπερ. Είναι δεν μου αφήνει καμία ε, κυρία, άμα θέλει να δώσω το λόγο πρώτα στον Νούτο, δεν έχω πρόβλημα. Νομίζω θα κάνουμε διαφορετικές ερωτήσεις εκείνος κι εγώ. Όλα τα μέτρα αυτά, τα οποία αποφασίστηκαν από τη Βουλή στην Ελλάδα, σίγουρα προϋποθέτουν μια διοίκηση η οποία να είναι σε θέση, παραδείγματος χάρη, να εισπράξει τους φόρους, να υλοποιήσει όλα αυτά τα μέτρα. Και αυτό που διαβάζουμε στον τύπο το γερμανικό είναι ότι τελικά υπάρχουν δύο διαφορετικές ε, φάσεις μεταξύ αυτών που αποφασίζονται και αυτών που υλοποιούνται και ότι συνεχίζουν να υπάρχουν ε, οφειλές οι οποίες αυξάνονται, ποσά τα οποία δεν πληρώνονται, η φοροεισπρακτική ικανότητα τελικά βλέπουμε να είναι κάπως ε, ε, αν θέλετε, η ίδια και ότι τελικά τα ποσά τα οποία χρειάζεται η Ελλάδα είναι εντυπωσιακά. Ε, ναι. Σε ό,τι αφορά ε, τους φόρους φόρων ή ε, τις άλλες υπερήμερες και λεξιπρόθεσμες οφειλές και την υστέρηση στη πρεξοφόρων. Όπως είπα και στην εισαγωγική μου ομιλία, υπάρχουν κάποια μέτρα για να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της ε, φορολογικής διοίκησης, της εφορίας και αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κάτι τέτοιο βέβαια προϋποθέτει και αποτελεσματική φοροεισπρακτική πολιτική και καθυστερημένων ε, φορολογικών οφειλών αλλά και των νέων. Αυτό αποτελεί τίμα του, του προγράμματος και ως προς την αιρεσιμότητα αλλά και ως προς την τεχνική συνδρομή που παρέχεται στην Ελλάδα για να βελτιωθεί η φοροσπρακτική ικανότητα της χώρας. Και στο θέμα της ε, βελτίωσης της φοροσπρακτικής ικανότητας ε, ε, επικεντρώνουμε σε μεγάλο βαθμό την τεχνική μας συνδρομή. Ο Μπουλμάν τώρα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ρομπέρτο. Εγώ πιστεύω ότι αδιαφυσβήτητα πρέπει να μπούμε σε έναν ενάρετο κύκλο και αυτό θα γίνει μόνο εάν συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα και οδηγηθούμε σε ένα σύγχρονο κράτος με κοινωνική δικαιοσύνη, και με σωστή κατανομή των βαρών. Από την άλλη, οι πιστωτές θα πρέπει να στηρίξουν δημοσιονομικά με τα πολιτικά μέτρα που προτείνουν και βεβαίως θα πρέπει να υλοποιηθούν οι αποφάσεις που ελήφθησαν πέρσι το καλοκαίρι για να δοθεί ε, λίγο οξυγόνο στην οικονομία. Χρειάζονται μέτρα που να οδηγούν σε ανάπτυξη, σε δημιουργία θέσεων απασχόληση. Οι αποφάσεις του Ιουλίου του 2015 αυτές καθεαυτές δεν θα τα δημιουργήσουν όλα αυτά. Χρειάζεται οξυγόνο, χρειάζεται ανάπτυξη και χρειάζονται αυτές οι τρεις φάσεις βέβαια που περιέγραψα για να φτάσουμε εκεί. Μέχρι το 2018 είναι πολύ ευαίσθητη χρονική περίοδος η πίεση επί της Νότιας Ευρώπης, των χωρών της Νότιας Ευρώπης θα συνεχίσουν με όλα αυτά τα μεταναστευτικά κύματα, τα κύματα των προσφύγων και γι' αυτό και χρειάζεται μια δίκαιη, κοινωνικά δίκαιη πολιτική. Η προτεραιότητα για την Ελλάδα βεβαίως είναι να ισχυροποιηθεί και να στηριχθεί η οικονομία, αλλά να μπορέσουν να παίξουν το ρόλο τους όλες οι κοινωνικές δυνάμεις. Και το θέμα της ε, διαχείρισης του χρέους που αναφέρατε, χωρίς ε, haircut, χωρίς ελάφρυνση, είναι δυνατόν να φέρει αποτέλεσμα. Μιλήσατε για διακυβέρνηση. Και πραγματικά αναρωτιέμαι μέχρι το 2018 που επαναλαμβάνω θα είναι μια πολύ ευαίσθητη χρονική περίοδος θα πρέπει κάτι να γίνει. Ε, βλέπουμε σήμερα να επανέρχονται θέματα εμπιστοσύνης και ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής ε, Κεντρικής Τράπεζας σίγουρα δεν είναι φίλος της ελληνικής κυβέρνησης αλλά προσπαθεί να κάνει κάποια πράγματα για να βοηθήσει αυτή την οικονομία. Αναρωτιέμαι λοιπόν, εάν αυτή η διαδικασία δεν φέρει τα επιθυμητά αποτέλεσμα, εάν δεν λειτουργήσει το σύστημα όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει, ο προληπτικός μηχανισμός νέων μέτρων θα ενεργοποιηθεί στην δεύτερη φάση και τελικά τι θα βελτιωθεί. Τι θα βελτιωθεί από αυτό έτσι όπως το έχετε προβλέψει. Καταρχήν ένα πολύ σημαντικό σημείο είναι ότι όλοι, όλα όσα κάνουμε, όλες οι αποφάσεις που λαμβάνουμε έχουν τον ίδιο στόχο. Γιατί ένα πρόγραμμα ε, δεν είναι αυτός σκοπός. Ούτε είναι αυτόματο δεν είναι το επίκεντρο των πάντων. Ένα πρόγραμμα, ένα μνημόνιο έχει ένα σκοπό. Επαναφορά στην ανάπτυξη, στις επενδύσεις, δημιουργία θέσεων απασχόληση και επιστροφή της Ελλάδας στις αγορέ. Και βρισκόμαστε σε μια σφαιρική διαδικασία. Και είναι η πρώτη φορά που μετά από χρόνια, σε ένα νυφάλιο κλίμα, αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα και το πρόβλημα των μεταρρυθμίσεων και το πρόβλημα του χρέους. Και πριν το 2012 είχε αναλυθεί η δέσμευση και επανελήφθη και πέρυσι και τώρα το κάνουμε. Και το μήνυμα που δίνουμε είναι ένα μήνυμα και προς τους επενδυτές και ένα μήνυμα και προς τις αγορές, ένα μήνυμα εμπιστοσύνης. Και όπως ρώτησε και πριν ο κύριος Μπάλτς, ζητούμενο είναι επαναφορά της ε, Οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα που την αναμένουμε για το δεύτερο εξάμεινο. Βέβαια, η ελληνική οικονομία έχει δείξει ότι είναι σε θέση να αντιδρά, να αντιδρά άμεσα και με έντονο τρόπο στα θετικά σημάδια. Γι' αυτό περιμένουμε να έχουν αποτέλεσμα. Τώρα για τη δεύτερη ερώτηση, για το ποιο. Ε, τώρα όταν έχουμε μεσοπρόθεσμα σενάρια, τα περισσότερα είναι πιθανολογίες. Αυτό που μετρά είναι να έχουμε ένα πραγματικό χάρτη πορεία, ένα φύλλο πορεία, ένα οδικό χάρτη. Και αυτό κάνουμε τώρα. Αυτό προσπαθούμε να διαμορφώσουμε, Ένα οδικό χάρτη για το χρέο και με τα μεσοπρόθεσμα μέτρα από το πρόγραμμα ε, και το θέμα του κουρέματος που είναι πιο μακροπρόθεσμο ζήτημα και που θα εξαρτηθεί από την επιτυχία των μέχρι τώρα δράσεων αλλά και από τη μακροπρόθεσμη προοπτική. Όλα αυτά θα διευκρινιστούν τις, τους επόμενους μήνες. Τώρα για το ποιο όλα αυτά θα ε, τύχουν ε, εξέτασης και παρακολούθηση στο πλαίσιο του Eurogroup που θα μείνει σε εγρήγορση και πολύ δραστήριο και ενεργό. Τώρα, αν θα έχουμε θεσμικές μεταρρυθμίσεις ε, για θέματα διακυβέρνησης της Ευρωζώνης, πα, και αυτό είναι πιθανό. Δεν ξέρω, είναι και ευκταίο κιόλα. Ε, γιατί καλό θα είναι να, περιλάβει, να περιλάβουμε και την δημοκρατική διάσταση και το θέμα του ελέγχου. Του ελέγχου μπορεί να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αποφάσεις που λαμβάνει το Eurogroup. Πάντω ε, σε αυτό το πλαίσιο, στο σημερινό πλαίσιο έχουμε παρακολούθηση του από το Eurogroup. Πάντως, στους επόμενους μήνες θέλουμε να διευκρινίσουμε τον οδικό χάρτη για το χρέος που πρέπει να είναι σφαιρικό, γενικός, πλήρης και θετικός γιατί εξαρτάται από το αν κανείς αισιόδοξο ή απεσιόδοξο όπως βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Πάντως από το τεχνικό επιτελείο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τη Διοίκηση έχουμε κάποια θετικά μηνύματα ότι μάλλον θα είναι θετική η έκβαση και εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί. Ο κύριος Κύρτσος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τους δύο επιτρόπους, τον κύριο Ντομπρόφσκης και τον κύριο Μοσκοβισή, γιατί ανεξάρτητα από το, την κυβέρνηση, την ελληνική, όποιος και να είναι, ε, έχουν βάλει μεγάλη προσπάθεια στο ελληνικό ζήτημα. Και νομίζω ότι το, ο Ιούνιος του 2016 είναι πολύ καλύτερος από τον Ιούνιο του 2015 που είχαμε μεγάλη αγωνία. Ε, θα ήθελα όμως να επισημάνω ορισμένα λεπτά σημεία που αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα, αλλά θα πρέπει κάποτε να αρχίσουμε να τα λύνουμε. Πρώτον, ε, με το σκεπτικό ότι πρέπει να λειτουργήσει ο ιδιωτικό τομέα καλύτερα στην Ελλάδα για να έχουμε ανάπτυξη και να μπορέσουμε να πάμε όλοι μαζί μπροστά. Το πρώτο που με ανισχύει είναι ότι δεν υπάρχει στρατηγική περιορισμού των non-performing loans, των κόκκινων δανείων που λέμε στην Ελλάδα. Είναι 45% του συνόλου, έχουν αυξητική τάση ε, αυτή τη στιγμή τα non-performing loans είναι στην Ελλάδα πάνω από 110 δισεκατομμύρια ε, και η η των τραπεζών είναι γύρω στα 130 δισεκατομμύρια. Είναι δηλαδή μια πολύ δύσκολη κατάσταση και παρά το γεγονός ότι σπάνια συμφωνώ με τον κύριο Μαριά, νομίζω ότι αν τα λεφτά και από τα S&P και από τα ANFAS τα λεφτά πέφτανε στο τραπεζικό σύστημα για να πέσουν στην πραγματική οικονομία, ίσως θα, ήταν καλύτερο το αποτέλεσμα από το να πέσουν στη μελλοντική διαχείριση του χρέους, γιατί πρέπει να, ανέβει η οικονομία. Το δεύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι η αύξηση της φορολογίας, η οποία για διάφορους κλάδους, όπως για παράδειγμα στον τουρισμό που είναι ανταγωνιστικός κλάδος στην Ελλάδα, είναι εντυπωσιακή. Δηλαδή ο ΦΠΑ VAT ε, πήγε από 13% στο 24% για εστιατόρια, ταβέρνες, όλα αυτά που προσφέρει η Ελλάδα. Επομένως, οι Ιρλανδοί μείωναν τη φορολογία στου τομεί που θέλουν να γίνουν ανταγωνιστικοί, εμεί τώρα αυξάνουμε τη φορολογία. Τώρα που θα οδηγήσει αυτό θα δούμε. Και το τρίτο που θέλω να σα επισημάνω, που έχει σχέση με το επιχειρηματικό κλίμα, είναι ότι υπάρχει ανοιχτή κρίση στο ε, δικαστικό και νομικό σύστημα στην Ελλάδα. Ε, judicial system, legal system. Ε, δηλαδή, έχουμε έξι μήνες απεργία των δικηγόρων, άρα δεν λειτουργούν τα δικαστήρια ε, γιατί οι δικηγόροι είναι σε αντίθεση με την κυβέρνηση, τους έχει, ασφαλίσει, τους έχει αυξήσει τη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές. Έχουμε δικαστές, ανώτατους δικαστές, που παίρνουν πίσω τα μέτρα, παίρνουν, δίνουν αυξήσεις σε αυτούς τους, δηλαδή δεν δέχονται μειώσεις μισθών ή συντάξεων, και το γενικεύουν κιόλα δημιουργώντα ε, ε, πρόβλημα και σε αυτήν και στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Άρα, πώς μπορείς να έχεις τώρα κλίμα εμπιστοσύνης με περισσότερους φόρους, ένα δικαστικό σύστημα που δεν λειτουργεί, και με κόκκινα δάνεια, non-performing loans στον ιδιωτικό τομέα που έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Αυτά τα πρακτικά ζητήματα πώς θα τα αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Uh, okay. On the question of... Ναι, όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια. Όντως, Πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα, το οποίο βεβαίως θα πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με τους ισολογισμούς των τραπεζών και βεβαίως θέλουμε να συνεχίσουν οι τράπεζες να δανείζουν και να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία. Πολλά μέτρα έχουν ήδη αποφασιστεί όπως παραδείγματος χάρη η αγορά για αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και βεβαίως ε, να δοθούν κίνητρα για αναδιάρθρωση του ε, τραπεζικού τομέα. Βεβαίως η ελληνική κυβέρνηση πήρε τα μέτρα που έπρεπε για το άνοιγμα των αγορών αυτών των μη εξυπηρετούμενων δανείων και σήμερα μπορούν οι τράπεζες να πουλήσουν σε μη τραπεζικούς οργανισμούς κάποια από αυτά, κάποιες κατηγορίες αυτών των δανείων. Και βεβαίως ε, η πώληση κάποιων τέτοιων ε, εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει αποφασιστεί και βεβαίως με μία εξαίρεση που είναι το ποσό των 140.000 ευρώ και εφόσον ένα τέτοιο δάνειο ε, έχει σαν υποθήκη την πρώτη κατοικία. Οι ελληνικές αρχές έχουν επίσης πάρει τις αποφάσεις τους όσον αφορά αυτές ε, τις ε, εταιρείες για την ε, αποπληρωμή αυτών των ε, οφειλών και βεβαίως ε, τις περιπτώσεις οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίων. Σκοπός μας είναι δηλαδή πραγματικά να στοχεύσουμε την καλύτερη υλοποίηση αυτών που έχουν αποφασιστεί, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για περιπτώσεις εξοδικαστικών διακανονισμών και Ξέρουμε ότι υπάρχουν ήδη κάποιες αποφάσεις ε, για τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά θα πρέπει και οι διαδικασίες πτωχεύσεων και ρύθμισης τέτοιων διαδικασιών να επιταχυνθούν και να αρχίσουν να λειτουργούν. Αυτό βεβαίως αποτελεί ε, τμήμα των συζητήσεων που λαμβάνουν χώρα, έτσι ώστε να μπορέσουν οι τράπεζες να ξαναρχίσουν να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Φάμπιο Μάση. Δύο σύντομες ερωτήσεις προς τον κύριο Μοσκοβισή. Γνωρίζουμε ότι στο επίκεντρο της κρίσης και πριν το δημοψήφισμα στην Ελλάδα, η ΕΚΤ αποφάσισε να μην δεχθεί ως, ε, παράγωγα, ως αγγίσεις ε, ε, ε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Και η θέση της ΕΚΤ ε, δικαιολογήθηκε με το, με το επιχείρημα ότι δεν έχει η Ελλάδα πρόσβαση στην σκεφαλαγορές, ε, ε, ότι έπρεπε να γίνει αποδοχή του προγράμματος. Τώρα έχει όμως γίνει αποδοχή του προγράμματος, οπότε υπάρχει περίπτωση να ξαναδεχθεί τα ελληνικά ομόλογα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί αυτό φημολογείται, μπορείτε να μας το επιβεβαιώσετε. Δεύτερον, στο Ταμείο Αποκαρατικοποιήσεων υπήρξαν κάποιες ενδείξεις ότι αν η Ελλάδα φτάσει ένα κατόφλι ιδιωτικοποίηση και ε, εσόδων από την ιδιωτικοποίηση, κάποια από τα κονδύλια αυτά θα χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις. Γιατί η Ελλάδα αυτό χρειάζεται, επενδύσεις. Γιατί η παραγωγικότητα είναι χαμηλή, οι επιχειρήσεις είναι μικρές και το κόστος του εργασιακού κόστους δεν επέτρεψε την ανάκαμψη. Οπότε χρειάζονται επενδύσεις. Οι επενδύσεις είναι κέρυες. Επίση δεν πήγαν και πολύ καλά αυτέ οι ιδιωτικοποιήσει. και αυτό δεν με ευνηδιάζει, δεν με εκπλήσει γιατί ε, με μια τέτοια οικονομική κατάσταση δύσκολα γίνονται επενδύσει. Οπότε χρειάζεται να δοθεί, να δοθεί όθηση στι επενδύσει. Αν όμω, ε, ε σε σχέση με τους στόχους αποκρατικοποίηση, ε, δύσκολα θα γίνει. Είπατε επίση ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί κάποιο είδου αναδιάρθρωσης χρέου. Νομίζω ότι Όλοι το γνωρίζουν αυτό. Ακόμη και ο κύριο Σόιμπλε, παρόλο που δεν θα το παραδέχονταν δημοσίω πολύ. Οπότε έχει αναβληθεί το θέμα μέχρι το 2018. Ε, φημολογείται ότι αυτό οφείλεται στις εκλογές, επικείμενες εκλογές στη Γερμανία. Γι' αυτό θέλετε, ήθελα να γίνει αναβολή μέχρι το 2018. Ο κύριος Μοσκοβισή, θέτε ερωτήσει για τι οποίε δεν μπορώ να σχολιάσω εκτενώς. Να σα απαντήσω πρώτα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Φυσικά δεν δικαιούται επίτροπος να σχολιάσει αποφάσεις ή μη αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πάντως ε, διάβασα τις ίδιες πληροφορίες με εσάς από ό,τι φαίνεται ότι το θέμα αναφέρθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και υπήρξε κάποιο θετικό κλίμα ότι θα μπορούσε να ξεπεραστεί το αδιέξοδο αρκεί να εφαρμοστούν κάποια προαπαιτούμενα. Δεν πρόκειται να το σχολιάσω, είπα. Πάντως αυτό κατάλαβα από την τελευταία συνέντευξη τύπου του Μάριο Ντράγκη, ότι μπορεί να ληφθούν κάποιες θετικέ αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα και από όλα τα θεσμικά όργανα. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως και ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχουμε στο Eurogroup και είμαστε από τους θεσμούς που έχουν συζητήσει με τις ελληνικές αρχές. Ας περιμένουμε λοιπόν. Κάποια θετικά σημάδια υπήρξαν. Θα δούμε αν θα ευοδοθούν περαιτέρω και αν, θα είναι, σωστή, αν είναι σωστή αυτή η ερμηνεία που δώσαμε. Σε ό,τι αφορά, σε το χρέος, εγώ δεν είμαι τόσο καλά εξοικειωμένο με τις εσωτερικές πολιτικές συζητήσεις στη Γερμανία όπω εσείς. Υπάρχουν κάποιοι νομικοί περιορισμοί όμως. Αυτό επαναλαμβάνει κυρίως ο Wolfgang Schäuble στο Eurogroup και ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές απαράβατες όπως ε, ότι δεν μπορεί να αλλάξει το μνημόνιο, το πρόγραμμα και ότι το, το κούρεμα είναι απάντηση. Πάντως υπήρξε μια η γενική συμφωνία σταδιακά να εγκύψουμε στα θέματα αυτά με βράχη, μέσο και μακροπρόθεσμες προσεγγίσεις. Και νομίζω ότι ως προς αυτό όλοι ακολουθούμε κοινή κατεύθυνση. Για το τελευταίο σας ερώτημα σας παραπέμπω ε, στο, στο μνημόνιο, στο, στην επιστολή του μνημονίου και στη συμφωνία του Αυγούστου είναι σαφές ότι το Ταμείο δεν είναι μόνο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, αλλά Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων και Επενδύσεων. Αυτό το σκοπό είχε από την αρχή. Και υπάρχει σαφή σύνδεσμος μεταξύ ε, της επιτυχίας ε, της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης ε, των εκταμιεύσεων των ταμείων και της τροφοδότησης των επενδύσεων. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν σεβαστά. Τώρα, τι θα επαναφέρει, θα επαναπροσελκύσει τις επενδύσεις προς την Ελλάδα μα η επιτυχία της όλης διαδικασία. Αυτό τα ξαναφέρει τι επενδύσει στην Ελλάδα και νομίζω ότι πραγματικά προσπαθούμε να στεφθεί με επιτυχία όλο, όλη αυτή η προσπάθεια για την Ελλάδα. Και στόχος του Eurogroup δεν είναι να αποφύγει ή να, να συζητήσει το πρόγραμμα ως αυτό σκοπό. Ο σκοπό του προγράμματο είναι να επαναφέρει τι ηθίκε και πρόσφορο έδαφο για τι επενδύσει. Και εξού και το, η δόση των 10,3 δις είναι ένα σημαντικό μήνυμα, χειρό μήνυμα προς την ελληνική οικονομία. Ότι η, γι' αυτό και οι μεταρρυθμίσει είναι τόσο απαραίτητες. Γι' αυτό και η συμφωνία που θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω είναι ένα μήνυμα προς τους επενδυτές. Αυτό καταλαβαίνουν οι επενδυτέ και οι αγορέ, ότι με τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων και με την ολοκλήρωση τη πρώτη αξιολόγηση, με την εκταμείευση και τη συνέχιση των προσπαθειών, ε, ενισχύεται η εμπιστοσύνη στην ικανότητα της Ελλάδας ε, να υιοθετήσει μεταρρυθμίσεις και να επανέλθει στον δρόμο της ανάπτυξης. Αυτή είναι η λογική της όλης πολιτικής ε, διαδικασίας που ακολουθούμε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ τους επιτρόπους, τον πρόψης και Μοσκοβισή. Εξαιρετικά χρήσιμη αυτή η συζήτηση, η και περιμένουμε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Όπως ξέρετε, στις 15 Ιουνίου θα υπάρξει μια συνάντηση, ένα workshop με ομιλητές από το Διεθνές Νομιστικό Ταμείο, την ε, Επιτροπή με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον Κλάους Ρέγκλινγκ. Θα μιλήσουμε για το θέμα του χρέους. Σας ευχαριστώ πολύ. Τέλος της συνεδρίασης.